Good morning to all of you. Καλημέρα σε όλους. Welcome to the budget. Καλώς ορίσατε στη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής ε, Budget 12 ε, Δεκεμβρίου. Υιοθετούμε πρώτα την ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχει μια ένσταση, κύριε Αντρέσεν, Όχι για την ημερήσια διάταξη. Είναι πρόβλημα που δεν βρίσκεται εδώ ο Επίτροπος ε, στην πρώτη συνάντηση μετά από την ε, εγκαθίδρυση της νέας επιτροπής. Τους έχουμε καλέσει. Θα έπρεπε να είναι εδώ και στη συνεδρία συντονιστών θα συζητήσουμε ε, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο έπρεπε να βρίσκεται εδώ. Να πείτε γι' αυτό κάτι τώρα ή αργότερα στην συνεδρία συντονιστών. Δεν είναι δυνατόν όταν έχουμε τόσο σημαντικές συζητήσεις όπως το Πολιτή δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να είναι εδώ. Θα σα δώσω πληροφορίε για το πότε θα έρθει ο κ. Χάρη στην Επιτροπή αργότερα. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Αν δεν υπάρχουν άλλε ενστάσεις, ε, συνεχίζουμε με τι ανακοινώσει του Πρόεδρου. Οι αποφάσει των συντονιστών τη 25 η Νοεμβρίου βρίσκονται στο φάκελο με τα έγγραφα τη συνεδρίαση και εδώ αν δεν υπάρχουν ενστάσεις θα θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί. Όπως ενημερωθήκατε μέσω email της γραμματείας στις 6 Δεκεμβρίου, επειδή το Συμβούλιο αποφάσισε να μην υιοθετήσει επίσημη θέση για το ΔΕΠ 5, δεν είναι δυνατόν η Επιτροπή Προπολογισμών εδώ του Κοινοβουλίου να υιοθετήσει επίσημη θέση για το ΔΕΠ 5. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι δεν θα ψηφίσουμε το ΔΕΠ 5 ούτε στην Επιτροπή μας, ούτε στην Ολομέλεια φέτος. Η άρνηση του Συμβουλίου να προχωρήσει σήμερα το ΔΕΠ θα περάσει. Δεν θα έχει εκτεθεί μέχρι το τέλος του 2019. Επίσης ενημερώθηκα από τη Φιλανδική Προεδρία ότι το Συμβούλιο σκοπεύει να υιοθετήσει τον κανονισμό του Συμβουλίου για τα μέτρα που αφορούν την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση του Γενικού Προπολογισμού της Ένωσης το 2020 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, με το Brexit δηλαδή, με διάφορες τεχνικές προσαρμογές ε, για να ληφθούν υπόψη οι απαραίτητες ε, τροποποιήσεις ε, στους κανονισμούς EGF και e USF μέχρι το τέλη του έτους αυτό. επειδή η Επιτροπή Προπολογισμών ψήφισε τη συνένεσή της για αυτό το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης λόγω του Brexit, Αυτέ οι προσαρμογέ είναι απαραίτητε μετά από διαβούλευση με την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Δεν απαιτείται περαιτέρω διαδικασία συνένεση. Αν δεν υπάρχουν άλλες αντιρρήσει όσον αφορά τα πρακτικά της συνεδρίαση της 25 η Νοεμβρίου, θα θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί. Πάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Πρώτα απ' όλα η σύναψη του πρωτοκόλου για την υλοποίηση τη ε, συμφωνία Εταιρική σχέση για ε, ε, την αλληλεία μεταξύ Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Δημοκρατία του Πράσινου Κροτηρίου. Ο φάκελο αυτό παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στη συνεδρίασή μα στι 25 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο. Δεν ξέρω, κυρία Μάρκε, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. <laughs> Uh, Καλημέρα, ο συνάδελφος μου ο Βαντόφσκι απάντησε ήδη, οπότε η απάντηση είναι όχι. Απλά να τονίσω ότι η έκθεση όπως επιβεβαιώνεται θα διαβιβαστεί ε, προς ψηφοφορία ε, είναι καλή αυτή η συμφωνία και για το πρασινοκροτήρι και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Τζόνσα, παρακαλώ, ένα λεπτό. Ξέχασα την κάρτα μου για να ψηφίσω, οπότε θα ψηφίσω ανατασχερός. Ωραία. Να σας υπενθυμίσω ότι πρόκειται για διαδικασία συνένεση, οπότε θα ψηφίσουμε ολόκληρη την γνωμοδότηση, οπότε περνάμε σε ονομαστική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. Everybody vote. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 18 υπέρ, 18 υπέρ ε, κατά δύο αποχές, ε, γιατί προσθέτουμε και την ψήφο. Δεν ήταν ισχυρός. Περνάμε στις ε, ε, μεταφορές στο τμήμα 3, κύριε Φεράντες. Α, για τα λοιπά τμήματα, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω εδώ τις ε, μεταφορές για το 4-2009 που μιλάει για δεσμεύσεις του λίματος 2001, εκμισθώσεις αγορές, ποσό 9.840.000 ευρώ για να χρηματοδοτήσουμε μια πρώτερη αγορά που έχει να κάνει με τη συντήρηση των κτηρίων και το δημοσιονομικό βάρος που σχετίζεται με μελλοντικέ πληρωμές. Δεν έχουμε μετάφραση. με τι εξοικονομήσει σε διάφορε δημοσιονομικέ ε, γραμμέ, ουδέτερη άποψη τώρα για την ΕΕΔ 2. 2019 άλλη μεταφορά για να ενισχύσουμε το λίμα 2100, τι σχετικές αγορές, πληροφορική και τεχνολογίες της πληροφορίας 2.447.000 καθώς και κρυπτογράφηση και απόρριτες πληροφορίες καθώς και τεχνολογία της επικοινωνίας 388.008 μετά παιδική σταθμή και παιδική φροντίδα 65.000 ευρώ, ε, λίμα 12.05 αποσπασμένοι στεγνωτικοί εμπειρογνώμονες 30.250 ευρώ και λίμα 1.500 κοινωνικές υπηρεσίες και υποστήριξη στο προσωπικό στους υπαλλήλους 14.900. Είναι σημαντικό για τη λειτουργία της ΕΕΔ η ενίσχυση του συστήματος τεχνολογίας και είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο προπολογισμό με τις δαπάνες για την πληροφορική που θα μπορέσουμε να αναθεωρήσουμε και θα μα επιτρέψει να αναθεωρήσουμε το αρχικό ποσό εφόσον χρειαστεί στο μέλλον. Έχουμε εξοικονομήσει από άλλε δημοσιονομικέ γραμμέ. Το έχουμε δει και με το διορθωτικό 5-2019 τη ΕΕΔ. Μπορούμε να ταμιεύσουμε τα ποσά αυτά για να καλύψουν αυτή τη δαπάνη. Επόμενο, επόμενη μεταφορά το 2019 για το Ευρωκοινοβούλιο. είναι 30.990.000 ευρώ για συντήρηση κτίριων ε, και μάλιστα για το Conrad Adenauer στο Λουξεμβούργο. Το ποσό αυτό είναι η παραδοσιακή άσκηση προσπάθεια συντήρησης και ανάκτησης ποσών, το ραμασάζ το λεγόμενο, των ε, ποσών του προπολογισμού, είναι εντός των κανόνων η διαδικασία αυτή και μας, επιτρέψει, μας επιτρέπει και μια ευελιξία. ο, το ποσοστό των ε, κονδυλίων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πριν από το ραμασάζ είναι 1,55 και αυτά έχουν να κάνουν και με τον προπολογισμό. Κάθε δημοσιονομική λοιπόν γραμμή πρέπει εδώ λοιπόν πρέπει να ασχοληθούμε ε, με αυτή τη δημοσιονομική διαδικασία και προτείνω να ψηφιστεί ε, και αυτή η μεταφορά και οι προηγούμενες δύο που σας υπέβαλα. What I propose to do is... Uh, λοιπόν, προτείνω πρώτα απ' όλα να ψηφίσουμε για τις πρώτες δύο μεταφορές και μετά την τρίτη. Και αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις, εάν συμφωνείτε, για το INF και το N2, δηλαδή την AED κύριε Άντερσεν, ναι, θα ψηφίσουμε διαφορετικά μεταξύ μας. Οπότε θέλουμε να έχουμε μια ψηφοφορία. Ωραία λοιπόν υποθέτουμε για τις πρώτες δύο, μάλλον θα υποθέταμε για τις πρώτες δύο ότι θα μπορούσαν να εγκριθούν, αλλά από ό,τι λέτε πρέπει να ψηφίσουμε για την κάθε μια ξεχωριστά. Υπάρχουν σχόλια για οποιαδήποτε από τις τρεις μεταφορές, γιατί πρέπει να ψηφίσουμε για τις τρεις ε, μεταφορές ξεχωριστά, πρέπει να ακούσουμε τώρα τα σχόλια σας. Κυρία Αρμό. Ναι, έχουμε επικεντρωθεί στο τρίτο, στην τρίτη μεταφορά. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε την κάθε μια από τι μεταφορέ, κατά αλλά για το τρίτο, για τη μεταφορά 30 εκατομμυρίων, ήθελα να μου πείτε από πότε ισχύει αυτό, γιατί η απόφαση τη Επιτροπή για αυτή την ανακαίνιση, αυτό το φρεσκάρισμα που μετά θα σχετιστεί με την πολιτική των κτηρίων, για το topping up λοιπόν, Πώς θα αλλάξει η απόφαση για το ρεμασάζ, εάν χρειαστεί. Πώς πρέπει να το αντιληφθώ και πώς θα μπορούσαμε να την αλλάξουμε αυτή την απόφαση. είναι 1,55% του προπολογισμού του Κοινοβουλίου, αλλά σε τι αναλογεί πραγματικά και πόσο χρόνο θα χρειαστεί για την πληρωμή αυτή. Υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα διαφάνεια στη δημοσιονομική διαδικασία, διότι καταλαβαίνω ότι επί χρόνια μιλάμε για μείον 5, μείον 7. Κάθε χρόνο υπολογίζουμε περισσότερα από ό,τι είχαμε στον προπολογισμό αρχικά. Κοιτάξτε, με τον σχέδιο προπολογισμού 5 κατάλαβα ότι τα 30 εκατομμύρια ήταν 45 εκατομμύρια εάν είχε περάσει το δευτικό 5. Ενώ τελικά τα 15 εκατομμύρια που ανακτήσαμε για τις πληρωμές, ε, δεν ξέρω αν έκανα λάθος, αλλά τα 15 εκατομμύρια ήταν απαραίτητα για τις πληρωμές για να καλύψουμε το κόστος του σεμιναρίου για τους βουλευτές, για τους ε, βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι λοιπόν σημαντικό όλα αυτά να τα δούμε από την αρχή. για να μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται με το ραμασάζ στο τέλος του κάθε, της κάθε χρονιάς. Λοιπόν, γιατί γίνεται αυτό το ραμασάζ, μου λέτε, είναι κάτι το οποίο έχει έννοια. Γιατί υπάρχει ο λεγόμενος πυρετός του, του Δεκεμβρίου. Δηλαδή όλοι όσοι έχουν ε, στα κονδύλια τους κάτι που τους έχει μείνει κάνουν ό,τι μπορούν τον Εύριο και τον Δεκέμβριο για να τα δαπανίσουν όλα. Γιατί αλλιώ θα τους κατηγορήσουν ότι δεν δαπάνησαν ε, τον προπολογισμό τους. Και πρόκειται για τομεί όπου για παράδειγμα αποφασίζουν οι βουλευτές μεμονωμένα αν θέλουν να κάνουν πλέον ταξίδια για να δαπανίσουν τον προϋπολογισμό τους. Αλλά πολλοί δεν το κάνουν. Άρα τα χρήματα αυτά μας μένουν. Τα χρήματα αυτά όμως θα έπρεπε τελικά να απαιτήσουν και περισσότερο κόστος. Πρέπει να πληρώνουμε για ό,τι δεν έχουμε δαπανίσει και τόκο. Γι' αυτό παρακαλέσαμε πάντα το Γενικό Γραμματέα στο τέλο να γίνεται αυτό το ραμασάζ, αυτή η συγκέντρωση πόρων από διάφορα σημεία για να πληρώνουμε τελικά, δαπανώντα περισσότερο για την αποπληρωμή λιγότερο τόκο για τα ε, χρέη μας, για τα κτίρια για παράδειγμα. Γι' αυτό προσπαθούμε ακριβώς να μειώσουμε παρόλα αυτά το ποσό το οποίο μένει για το ραμασάζ. Παλιά ήταν 100-120 εκατομμύρια. Τώρα έχουμε πέσει στα 40. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα μειώσουμε. Αλλά ε, έχει έννοια. Πάντα κάτι θα μείνει. Δεν είναι δυνατόν ακριβώ να προγραμματίσει, να ξοδέψει και το τελευταίο ευρώ τα ταξίδια που έχουν προγραμματίσει οι βουλευτές μπορεί να αλλάξουν. Δεν θέλουμε λοιπόν να τα ε, χάσουμε. Καλύτερα να, αυτά τα χρήματα που μένουν να τα πληρώσουμε, να πληρώσουμε περισσότερο για να πληρωμή το χρόνο μας για τα κτίρια για παράδειγμα για να πληρώσουμε λιγότερους τόκους. Αυτή είναι η έννοια του Ραμασάζ. Η κυρία Γαρδιαθάβαλ. Ευχαριστώ. Ναι, αυτό το Ραμασάζ αυτή η μεταφορά σκούπα πάντα προκαλεί συζητήσεις. Υπάρχουν δύο τρόποι να το δεις. Το είπε και η κυρία Χολμάιερ για χρόνια. Το μασάζ, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή πολύ μεγαλύτερο ποσό μεταφέρονταν με το ραμασάζ. Γι' αυτό εμείς είπαμε ότι πρέπει να μην υπολογίζουν περισσότερα από όσα θα ξοδέψουν για ορισμένες γραμμές του προπολογισμού και καταλαβαίναμε βέβαια ότι ορισμένοι το κάνανε επίτηδες για να έχουν περισσότερα χρήματα. 30 εκατομμύρια για τη χρονιά που συζητάμε δεν είναι και τόσο κακό ποσό. Έχουμε βελτιώσει την κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να, να βλέπουμε και τα επόμενα χρόνια ποιε γραμμέ του προπολογισμού υποεκτελούνται για να μειώσουμε περισσότερο αυτό το ραμασάζ. Αυτά γενικά για το ραμασάζ. Τώρα για αυτό το ποσό του ραμασάζ να το αξιοποιήσουμε για την αποπληρωμή των χρεών για τα κτίρια είναι η καλύτερη δυνατότητα. Διότι βεβαίω με 30 εκατομμύρια πολλά μπορούμε να κάνουμε. Αλλά στι 10 και 12 Δεκεμβρίου δεν νομίζω ότι θα ήμασταν σε θέση να βρούμε προγράμματα, να τα χρηματοδοτήσουμε σωστά για να αξιοποιήσουμε αυτά τα 30 εκατομμύρια. Το CAD, το κτίριο Contra Dandenau στο Λουξεμβούργο, είναι πίθο των Δαναίδων, εντάξει. Αλλά, εν πάση έχει χτιστεί τώρα, υπάρχει ένα σχέδιο αποπληρωμής του χρέους για το κάτι και θα το βελτιώσουμε έτσι. Τώρα, το να ζητάμε επίσης να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για να καλύψουμε το κόστος του Brexit είναι ένα θέμα περισσότερο φιλοσοφικό παρά λογιστικό. Εάν μείνουν οι ευρωβουλευτές και αν μείνουν οι βοηθοί και αν πρέπει να πληρώσουμε όλα τα έξοδα, όλες τις δαπάνες, θα πρέπει να τροποποιήσουμε τον προπολογισμό. Δεν είναι πολιτικό θέμα αυτό, είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Γι' αυτό πρέπει να τροποποιήσουμε τον προπολογισμό. Γιατί αν δεν το κάνουμε, τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Δεν ξέρω αν θα έχουμε άλλο κάποιο Brexit ή για κάποιο άλλο λόγο πρέπει να τροποποιήσουμε τον προπολογισμό. Μπορούν να μα πούνε, όχι, όχι, όχι, έχετε αρκετά λεφτά, κάντε κάποιε προσαρμογέ εσωτερικέ. Όπω έχει υποθεί στο παρελθόν. Αυτό θα σήμαινε ότι δεν έχουμε κανένα περιθώριο μετά. Δεν θα είχαμε κανένα περιθώριο μετά για να μειώσουμε, για παράδειγμα, τα ενυπόθηκα δάνειά μας. Είναι λοιπόν θέμα αυτού αρχής. Δεν είναι θέμα ότι θα μπορούσαμε να βρούμε 15 εκατομμύρια τώρα, αλλά για να μην να προλάβουμε μελλοντικέ παρόμοιε συζητήσει αν προκύψει παρόμοια ανάγκη. Γι' αυτό ζητάμε από την Επιτροπή να τροποποιήσει τον προπολογισμό μας για να πληρώσουμε για τον Brexit. Να μην το ξεχάσουμε αυτό. Και αν μείνει αλλού κάποιο ποσό, μπορούμε να συζητήσουμε για το πώς θα το δαπανίσουμε. Αλλά τώρα στο σημείο που βρισκόμαστε, νομίζω το πιο εύκολο είναι να προκαταβάλουμε κάποιες δόσεις από τον υπόθηκο δάνειό μας. Αυτά. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Η DG Fins μήπως μπορεί να μας εξηγήσει λίγο καλύτερα τι γίνεται με αυτό το κτίριο Κόντρα Adenauer στο Λουξεμβούργο. Είναι εδώ ο κύριος Κλετή ή ο κύριος Μπάς. Δεν είναι εδώ. Να σας δώσω κάποιες εξηγήσεις εγώ. Το CAD, το κτίριο Κόντραντ Αντενάουερ, ξεκίνησε εδώ και χρόνια και προχωράει, κοντεύει να ολοκληρωθεί. Θα δείτε το συνολικό κόστος εδώ στον πίνακα. Είναι 469 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε χρηματοδοτήσει βεβαίως την κατασκευή με τρόπο τέτοιο που μας πήραν, μας έδωσαν διάφορες τράπεζες δάνεια κατά τη διάρκεια της ε, κατασκευής θυμίζω ότι όλη αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε όταν ακόμη οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν μπορούσαν να ε, ζητήσουν απευθείας δάνεια από τράπεζες. Αυτό ξεκίνησε μόνο με τον ε, δημοσιονομικό κανονισμό όπως τροποποιήθηκε το 2012. Από τότε και μόνο μπορούμε να πάρουμε απευθείας δάνεια από τράπεζες. Αυτό όμως που με συνέπεια κάνουμε τα τελευταία χρόνια είναι μέσω του ραμασάζ τα οποία ραμασάζ οι πόροι δηλαδή από το ραμασάζ χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς όπως για παράδειγμα τα γραφεία σύνδεση κτλ αλλά γενικώ αξιοποιούνται και για αυτήν την αποπληρωμή των ε, κτηρίων. Για παράδειγμα, ένα τμήμα αυτού του ραμασάζ χρησιμοποιείται όμως και για πληροφορική. Δεν είναι δηλαδή ότι όλοι οι πόροι το ραμασάζ πάνε στα κτίρια. Ωστόσο, να επανέλθω στα ραμασάζ των τελευταίων ετών. Μας έχουν επιτρέψει να φτάσουμε τώρα σε τέτοια κατάσταση που έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο όπου το συνολικό κόστος του κτηρίου έχει σχεδόν πλήρως καλυφθεί. Χρειαζόμαστε μόνο 72 και με αυτά τα 30, λοιπόν, θα, συγγνώμη, 74 χρειαζόμαστε ακόμη και με αυτά τα 30 θα πέσουμε στα 44. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους ε, είναι σκόπιμο είναι ότι έχουμε μειώσει τους τόκους κατά 4 εκατομμύρια Ξέρετε ότι αν έχει ζητήσει κειμενόμενο επιτόκιο, αλλάζει και δεν ξέρεις πόσο θα χρειαστεί να πληρώσεις. Οπότε δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς θα, πόσο ακριβώς θα εξοικονομήσουμε, αλλά θα είναι τουλάχιστον 4 εκατομμύρια. Λιγότερους στόχους λοιπόν. Και αυτό επίσης έχει το πλεονέκτημα ότι η αποπληρωμή δεν χρειάζεται να γίνει απευθείας από τον προπολογισμό του επόμενου έτους είναι πρόορες πληρωμές και θα έχουμε πλήρη κατοχή του κτηρίου νωρίτερα επειδή η καιρή είναι αβέβαιη έχουμε τον Brexit η διαπραγματεύση για το νέο πολίτες πλαίσιο είναι ακόμη σε εξέλιξη δεν ξέρω εάν ε, οι προτάσεις μας θα γίνουν δεκτές αλλά δεν θεωρώ ότι στο κεφάλαιο 7 θα υπάρξουν μεγάλες αυξήσεις τα επόμενα χρόνια οπότε οι νωρίτερε πληρωμέ σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι θα γίνουμε πλήρη, κύριοι του κτηρίου μας νωρίτερα. Σε αβέβαιους καιρούς αυτό είναι θετικό. Γι' αυτό ακριβώς υποβάλαμε το αίτημα αυτό για μεταφορά πιστώσεων. Γιατί θεωρούμε ότι είναι χρηστή διαχείριση. Ό,τι σου περισσέψει να το αξιοποιήσεις για να πληρώσεις λιγότερους τόκους. Καλύτερα αυτό παρά να πει στου διατάκτε ε, ε έχουν μείνει κάτι λεφτά, κάντε τα ό,τι θέλετε. Είπα είναι αβέβαιοι καιροί. Έχουμε το DAB, το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού 5. Και αυτό το πλεόνασμα, αντί να προβλέπουμε έλλειμμα, είναι καθυσχαστικό. Δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση πριν το πέρα τη εκλογική διαδικασίας. Δεν ξέραμε ακριβώς τι θα γίνει, πόσοι βουλευτέ θα είναι τελικά. Γιατί το Brexit, το οποίο συνεχώς μετακινείται, βέβαια κάνει πολύ δύσκολη την προσπάθεια υπολογισμού. Επίσης, αυτό που μας ενδιαφέρει, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο, είναι πόσοι επανεκλέγονται. Γιατί όσο περισσότεροι επανεκλέγονται, τόσο περισσότερο, συγγνώμη, όσο λιγότερο επανεκλέγονται, τόσο μεγαλύτερα είναι τα έξοδα γιατί οι καινούργοι βουλευτέ έχουν να κάνουν περισσότερε προσαρμογέ, παίρνουν περισσότερο χρόνο για να προσλάβουν του βοηθού του και δεν ξέρουμε πόσα θα χρειαστεί να δαπανίσουμε πότε. Οπότε αυτό μπορεί τελικά, επειδή καθυστερούν να προσλάβουν, όπω είπα, το προσωπικό του νέοι βουλευτέ, σημαίνει ότι μα μένει πλεόνασμα. Το ραμασάζ τον Οκτώβριο ήταν στο 3,1. θα είπε 2% ότι θα είναι τελικά. Και γι' αυτό χρειάστηκε να κάνουμε αυτό το DAB 5. Αν δεν το κάναμε όμως αυτό, αν δεν είχαμε προβλέψει, εάν δεν είχαμε κάνει τις αναγκαίες δαπάνες, τότε η μάζα των 70 ε, εκατομμυρίων που είναι οι δαπάνε για τους μισθούς του προσωπικού μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί. Ο ΝΤΑ 5 δεν χρειάστηκε. Αλλά το χρειαζόμασταν τον Απρίλιο, θεωρούσαμε ότι το χρειαζόμασταν όταν το ζητήσαμε. Όταν έγινε η πρώτη αναβολή του Brexit, από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο, τότε χρειάστηκε να αδειάσουμε πλήρως το αποθεματικό έκτακτης ανάγκης που είχαμε ζητήσει. Και είχαμε και ένα πρόβλημα με την πολιτική, την επικοινωνιακή, γιατί είχαμε μεγάλες δαπάνες ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο για, τον, ε, για την εκλογική διαδικασία. Ήταν κάτι που δεν είχαμε προβλέψει. Τον Απρίλιο, που θεωρούσαμε ότι θα είχαμε έλλειμμα, εάν ο, πρό, ο πρόεδρος, με κύριε Μπάς. Σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες αυτές. Καταλάβαμε, πιστεύω, μέσα σ' άκρες, πρέπει να πρόκειται για να συνοψίσω, αν σας κατάλαβα καλά, σε σχέση με αυτό το ραμασάζ θα χρειαστείτε 40 εκατομμύρια επιπλέον στο μέλλον. Αυτό είναι σωστό. Ναι, σωστά το λέτε. Αυτό συμπερασματικά. Και αυτό είναι συνέπεια του γεγονότος ότι το 2012 επιλέξατε ε, ένα δάνειο σταθερού επιτοκίου, το οποίο είναι κατανοητό ότι κάνατε αυτό το πράγμα τότε, το οποίο σημαίνει τότε ότι δεν γνωρίζετε τα μυστικά, δεν ήσασταν στο και στο κύκλο του κύριου Ντράγκη. Αυτό είναι καλό, αστείευομαι. Αλλά ήταν απόλυτο κατανοητό το 2012 να επιλέξετε ένα σταθερό επιτόκιο. Αυτό μας εξηγεί επαρκώς την κατάσταση. Το παρά όπως ζήτησε ο κ. Αντρέσεν θα ψηφίσουμε ξεχωριστά για τα τρία ζητήματα. Πρώτον, για το INF 4219 του δικαστηρίου άρχιδη ψηφοφορία ψήφισαν άπαντες πέρας ψηφοφορίας 21 υπέρ και δύο εποχές πάμε στο 1.2 κάθετος 2019 της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης άρχεται ψηφοφορία Ψήφισαν άπαντε. Πέρας ψηφοφορία. 19 υπέρ, 1 κατά και 3 αποχές. Και τέλος μεταφορά C19 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάθετος 2019. C19 κάθετος 2019. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας ψηφοφορίας. 12 υπέρ, 3 κατά, 8 αποχές. Εγκρίνονται και τα τρία. Ευχαριστούμε. With respect to building policies. Όσον αφορά την πολιτική για τα κτίρια, Πρώτα απ' όλα το κτίριο Στέφαν Τσβάικ, το κέντρο επισκεπτών. Δίνω το λόγο στην κυρία Αγία, αφού η κυρία Κέλλερ δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ σήμερα. Κυρία Αγία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι η Φαμπιέν Κέλλερ δεν μπορούσε να είναι εδώ. Θα την εκπροσωπήσω εγώ όσον αφορά την πρώτη ψηφοφορία για το Κέντρο Επισκεπτών της ΒΑΕΚ, το σχέδιο που προτείνει το Κοινοβούλιο συνίσταται στη δημιουργία ενό νέου χώρου υποδοχή επισκεπτών στο ε, κτίριο της ΒΑΕΚ. Ε, ε, Σκοπό είναι να δημιουργηθεί μια νέα αίθουσα σεμιναρίων πέραν αυτών που υπάρχουν στο ΣΠΑΚ για να υποδεχόμαστε περισσότερου επισκέπτε και έτσι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να υποδεχόμαστε επισκέπτε και κατά τη διάρκεια των εργασιών στο κτίριο Σπακ λίγο πάνω από 10 εκατομμύρια θα στοιχήσει και θα χρηματοδοτηθεί από τη γραμμή 2007 για τρία χρόνια. Μέχρι το 2021 οι εργασίες θα ξεκινήσουν το 2020 για να ανοίξει το κέντρο στις αρχές του 2022. Η, η άποψή μας είναι ευνοϊκή. Υπάρχει κάποιο σκιώδης που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Αν όχι, πάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 3 κατά. Εγκρίθηκε. Το επόμενο σημείο αφορά το κτίριο Μπέλμο, αφορά τις, ε, ε, την ενοικίαση ε, γραφειακών χώρων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας ε, παρουσιάσω την ανάλυση της κυρίας Κέλλερ για το κτίριο Belmont. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, Εξωτερικής Δράσης θέλει για 15 χρόνια να έχει τη χρησικτησία αυτού του κτίριου ε, Belmont. Στόχος είναι να αυξηθεί ο γραφειακός χώρος ώστε να αντιμετωπιστεί η αύξηση προσωπικού και η σημερινή και αυτή που προβλέπεται από το 2021 θα αντικαταστήσει δύο άλλα κτίρια που ενοικιάζει η υπηρεσία αυτή, το Μπελιακατό και το Μερόντο, που είχαν ξεκινήσει το 2018 και το 2017 αντίστοιχα. Πρέπει να γίνουν κάποιε εργασίε για να προσαρμοστεί απόλυτα στις νέε χρήσει. Έτσι, το κτίριο θα μπορούσε να είναι έτοιμο τον Οκτώβριο του 2020. Αυτό το νέο συμβόλαιο θα βοηθήσει να αυξήσουμε την επιφάνεια κατά 7.500 τετραγωνικά μέτρα σε σχέση με, ε, με το σημερινό εμβαδόν λίγο πάνω από 4 εκατομμύρια το σημερινό κόστος ετησίως μαζί με τα εργασίες συντήρησης ε, και το ενίκιο και τους λόγους τις δαπάνες. Από τα κεφάλαια 200-201 ε, των κονδύλων για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ωστόσο θα χρησιμοποιηθούν και επιπλέον μεταφορές και έτσι θα κινητοποιηθούν τα απαραίτητα ποσά με παρακαθορισμό των προτεραιοτήτων Παρ' όλα αυτά, εμεί έχουμε επιφυλάξει όσον αφορά τον Πελιαρεκατό, ένα κτίριο το οποίο θα αντικατασταθεί από τον Πελμό και η ενοικίαση του οποίου το 2018, είχε ξεκίνησε μόλι το 2018 και που μπορεί να ολοκληρωθεί ε, μέχρι το 2023, εκτό ε, αν κάποιο άλλο οργανισμό ε, πάρει το συμβόλαιο ενοικίαση. Δεν υπάρχει όμω κάποια γραπτή εγγύηση γι' αυτό. Έχουμε λοιπόν ευνοϊκή γνώμη, ωστόσο θα θέλαμε να δοθούν εγγύησει για την ε, ε, διαβίβαση του ε, συμβολέου νοικιάσης του Μπελιαρέκατο. 100. Δεν ξέρω αν θα μπορούσατε να μας δώσετε παραπάνω πληροφορίες. Mr. Larson, yes, please. Ο κύριος Λάρσεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τι συγκεκριμένε ερωτήσει, για τι εγγυήσει, για το Μπελιάρ 100 και ποιο μπορεί να αναλάβει το κτίριο αυτό. Εμείς δεν μπορούσαμε να δώσουμε η ΕΕΔ ε, εκδήλωσε ε, το ενδιαφέρον της γιατί εμείς δεν αναλάβαμε Ε, εμείς λοιπόν αναλάβαμε για αυτό το λόγο και η εγγύηση δεν μπορεί να είναι επίσημη αυτή τη στιγμή, όμως ευχαρίστως να σας αποστείλουμε και γραπτός εγγύησης. Εξ αρχής δεν ξέρω ε, γιατί επιμένουν και ποιες είναι οι ανάγκες τους ακριβώς, αλλά φαίνεται ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Άλλοι σκιώδεις εισηγητές, κυρία Χολμάγερ. Έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις για την... Ε, διότι είναι διπλάσια η επιφάνεια από αυτή που έχει τόσο τώρα στο κτίριο αυτό. Ο διπλασιασμός σημαίνει ότι θα αλλάξει και κατανομή του προσωπικού θα ανέβει ο αριθμός. Εδώ λοιπόν είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε και από την προοπτική του προπολογισμού ότι έχουμε περισσότερα για τους αποσπασμένους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και τελικά το προσωπικό που είναι διορισμένο δεν ε, αυξάνεται. Δηλαδή τελικά χρηματοδοτούμε διακυβερνητικές δομές και προσωπικό μέσω από την ε, πολιτική των κτηρίων. Ελπίζω να έγινε κατανοητό αυτό που λέω. Και το δεύτερο είναι ότι καλό θα, είχε, πρέπει, καλό θα ήταν να έχουμε και ε, μια εικόνα για τη μεσοπρόθεσμη προοπτική των εργασιών της ΕΕΔ πώς προβλέπετε να εξελιχθούν τα πράγματα. Διότι μέσα σε τρία χρόνια έχουμε αλλαγή κτηρίων, κάτι που δεν είναι πάρα πολύ καλό για το πώς διαχειριζόμαστε το κόστος λειτουργίας. Ε, κάποια κτίρια, κάποιων κτίριων μάλλον λίγη το μισθωτήριο το 2021 και παραπέρα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε εάν μπορούμε να κάνουμε εκεί κάτι και μετά για την ΕΕΔ μπορεί ε, το Κοινοβούλιο να κάνει κάτι με τα γραφεία των προσωπιών ε, γιατί ξέρετε ότι και από εκεί υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες. Έχετε ένα ωραίο μεγάλο κτίριο, αλλά και το, το κοινοβούλιο θα ήθελε να οργανώσει τις υποδομές του διαφορετικά σε διάφορες χώρες Δεν ξέρω αν μπορείτε να απαντήσετε και στις τρεις ερωτήσεις, αλλά η δεύτερη κάπως απαντήθηκε, μάλλον η πρώτη απαντήθηκε κάπως από τη δεύτερη από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή το τι θα κάνουμε με την πώληση κτηρίων την εκμίστοση ε, μπορεί να γίνει από τη διαδικασία του προπολογισμού. Αλλά θα πρέπει και κάπως να συμφωνήσουμε για τη διαχείριση των Κύριε Λάρσον, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χόλμαγερ, ξέρω ότι είστε γνώστρια της κατάστασης και όχι μόνο για την πολιτική των κτηρίων. Για την αύξηση του προσωπικού, το πρώτο που ρωτήσατε. Ο σκοπός μας δεν είναι απλώς να το κάνουμε για πλάκα. Είναι υπερπλήρες το κτίριο έχουμε εγκατασταθεί σε τέσσερις διαφορετικά σημεία και μόλις την περασμένη εβδομάδα προβλέπαμε αύξηση προσωπικού 169 άτομα το 2020. 112 θα είναι στα κεντρικά. Σε ό,τι με αφορά, μπορούμε να υπολογίσουμε ποιοι είναι ταμπορέ, ποιοι είναι μόνιμοι, ποιοι είναι αποσπασμένοι. Έχουμε διαφορετικές κατηγορίες στα διάφορα γραφεία. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι κάποιοι θα πρέπει να δουλεύουν διαφορετικά από άλλους, δηλαδή με τους διατοτικούς που έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση για την αποσπασμένη εθνική εμπειρογνώμονες. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι ε, στη διάθεσή μας. Είναι διαφορετική η συζήτηση. Έχουμε ε, το 2020 θα έχουμε διαφορετικό, διαφορετική αύξηση του προσωπικού. Ευχαριστούμε γενικώ το Κοινοβούλιο για την ε, σημαντική αύξηση. Είχαμε και την προηγούμενη διετία μια ξαφνική αύξηση. Έχουμε επίση και την στρατιωτική και πολιτική διάσταση, όπω τη λέμε, αυτού που αναλαμβάνουν την ελοπίση ε, των αποστολών μα στο εξωτερικό. Είναι δύο τομεί που αναπτύσσονται ταυτόχρονα πολύ γρήγορα δεν είναι αλήθεια ότι θα είναι μισογεμάτο το κτίριο. Θα είναι υπερπλήρε από την αρχή. Και το συζήτησαμε με του εισηγητέ. Λένε ότι είναι κρίμα να έχουμε αυτή την κοτόφθαλμη θεώρηση, διότι αν αυτή η τάση συνεχιστεί στην ίδια κατεύθυνση, σε μια διετία θα πρέπει να ξανάρθω και να σα ζητήσω κι άλλα από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, Κάναμε όσο χώρο μπορούσαμε, ε, στριμωχτήκαμε, γιατί έχουμε ένα μεγάλο κτίριο, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, μπορούμε να ε, στριμωχτούμε κι άλλο, αλλά Έχουμε μια καλή τιμή τώρα που μας προσφέρεται. Πρέπει να το κάνουμε γιατί είναι έξυπνο. Ε, και η τιμή είναι σε καλά επίπεδα για την αγορά. Είναι ανταγωνιστική. Ε, είναι και για μας και για εσάς ενδιαφέρον. Για ένα μικρό διάστημα τουλάχιστον μέσω πρόθεσμα μπορούμε να οργανωθούμε σε τρία βασικά κτίρια. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Τρία. Ε, διότι εκεί που βρισκόμαστε τώρα που ξέρετε χτίζουμε ένα καινούριο που είναι σε μια ιδιαίτερα ασφαλή περίμετρο. Οπότε ερπίζουμε ότι θα έχουμε διοικητικά μια προστατευμένη περιοχή για να μην έχουμε περισσότερα ε, έξοδα και κόστος για την ασφάλεια. Και το τρίτο, από την άποψη των κτηρίων, ήταν μεγάλη κανένα πρόβλημα να έχουμε τουλάχιστον 140 ε, συγκατοικήσεις, ε, μισθώσεις από κοινού. Ε, δεν μας ενόχλησε καθόλου. Δεν ενισχύει λοιπόν ότι δεν τα βρίσκουμε με τα άλλα θεσμικά όργανα όταν υπάρχει διάθεση συνεργασία. Υπήρξε μια υπόθεση, μπορεί να συμβεί αυτό. Κάποιε φορέ είμαστε υπερπλήρει και δεν μπορούμε να πάρουμε άλλου. Αλλά Κάποιε φορέ υπάρχουν πολιτικοί λόγοι. Δεν είναι βεβαίω η δική μου αρμοδιότητα για να το πω, αλλά τα προβλήματα ε, προκύπτουν για άλλου λόγου. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την ε, κουβέντα, αλλά ευχαρίστω να δεχτούμε κόσμο από άλλα θεσμικά όργανα, από τα κράτη-μέλη. Το 7% των αντιπροσωπιών μα, το 7% τη επιφάνειά μα ε, είναι κατηλημένο από άλλου, όχι από εμά. Ευχαριστώ, κυρία Χόλμαερ. Κοιτάξτε. Το 7% είναι σε μεγάλο βαθμό άλλες πρεσβείες. Ρώτησα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι ακριβώς ε, καλύπτει, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη η γενοδορία έναντι του Κοινοβουλίου. Εάν ε, προβλέπονται νέα κτίρια, θα ήταν καλό η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση να ρωτήσει το Κοινοβούλιο για να συμπεριληφθεί στον σχεδιασμό για τα νέα κτίρια. Και θα πληρώσουμε ό,τι μα αναλογεί. Όπω γίνεται και για άλλα γραφεία μα. Για τα άλλα γραφεία μα, βεβαίω, έχει υπάρξει γενοδορία του Κοινοβουλίου. Και για το πρώτο σημείο. Οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονε θα πρέπει να δούμε ακριβώ πόσοι είναι διότι στην ουσία έτσι τα κράτη-μέλη δημιουργούν διακυβερνητικές δομές τις οποίες δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Και το Κοινοβούλιο, συγγνώμη μάλλον καλύτερα το Συμβούλιο, στην ουσία θέλει να μειωθεί το προσωπικό της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου και να αυξηθεί ο αριθμός των ε, εθνικών εμπειρογνωμόνων τους οποίους δεν έχουμε καμία δυνατότητα να ελέγξουμε. Συνεργάζονται μαζί μας ε, αν θέλουν, αλλά αν τα κράτη-μέλη τους που να μην συνεργάζονται ή να φύγουν, έχουν ε, κάθε εξουσία να το κάνουν. Και στην ουσία μειώνεται η δυνατότητα του Κοινοβουλίου να συνεργαστεί με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Και αυτό ισχύει και για άλλους οργανισμούς. Αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα που πρέπει να το δούμε. Κατά τα άλλα μπορώ να συμφωνήσω. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Θέλει κανείς ε, άλλος κοιόδης να παρέμβει, να σχολιάσει. Όχι. Να ψηφίσουμε. Ηλεκτρονικά άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 16 υπέρ, 3 κατά, 5 αποχές. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία των ψηφοφοριών. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, κτηριακή πολιτική και πάλι. Τα γραφεία μας στο ε, Πεκίνο. Παρακαλώ κυρία Αγέ και εδώ και πάλι εκπροσωπώ την Φαμπιέν Κέλλα. Λοιπόν, για το θέμα αυτό, ανανέωση της μίσθωσης για τα γραφεία της Ένωσης στο Πεκίνο. Περί τίνος πρόκειται. Ανανέωση της μίσθωσης. Δεν χρειάζεται να περάσει από την ε, αρχή επί του προπολογισμού συνήθως τέτοιο θέμα, αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η μίσθωση αυτή, η νέα δηλαδή, σημαίνει αύξηση 20% του μισθώματος. Περιμένουμε να υπάρξει ένα ενίο κτίριο για να ε, φιλοξενήσει όλη την ε, υπηρεσία που τώρα είναι την αντιπροσωπεία μας που τώρα είναι σε δύο κτίρια και η, το μίστομα δεν έχει αυξηθεί από το 2002 οπότε αυτή η αύξηση του 20% εκπροσωπεί όλη αυτή την περίοδο λοιπόν πρώτη ερώτηση ποιο θα είναι το ποσό του ενοικίου μετά την αύξηση και εδώ μας λέτε ότι θα είναι για τέσσερα χρόνια αυτό το νέο ενίκιο. Και είπατε ότι το κτίριο που θέλουμε να χτίσουμε θα πάρει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια. Γιατί να μην προβλέψουμε λοιπόν ε, μια μίσθωση πέντε ετών για να καλύψουμε δεχόμενη καθυστέρηση στην οικοδόμηση του νέου κτιρίου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Για άλλου η κυρία Χολμάια. Κοιτάξτε, έχω πολύ διάθεση να είμαι μαχητική σήμερα. για το κτίριο αυτό. Συμφωνώ σήμερα, αλλά θα απορρίπτω από πλευρά του ΕΛΚ οποιαδήποτε παρόμοια προσπάθεια στο μέλλον, αν δεν υπάρχει πλήρη συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Η κυρία Γουρδιαθάβαλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση. Όταν υπογράψαμε το προηγούμενο συμβόλαιο και πότε ακριβώς ήταν Τώρα ξέρουμε ότι πρέπει να περιμένουμε τέσσερα χρόνια τουλάχιστον πριν περάσουμε στο νέο κτίριο για να ολοκληρωθεί η οικοδόμηση του δεύτερου τμήματος του νέου κτίριου και εντωμεταξύ βεβαίως ε, θα ανέβει το ενίκιο. Ακόμη και 60% αν μας πρότεινε αύξηση θα το δεχόμασταν διότι δεν έχουμε άλλη λύση. Και δεν ξέρω. Δεν μπορούσαμε να έχουμε προβλέψει νωρίτερα ότι θα χρειαζόμασταν περισσότερο χρόνο στο παλιό κτίριο μέχρι να ολοκληρωθεί το νέο για να μπορέσουμε να τα κομίσουμε. Ευχαριστώ, όλοι ο Πρόεδρος. Ο κύριος Αντρέισεν. Ναι, και εμείς είμαστε υπέρ, αλλά έχω ρωτήσει, όπως και η Άιντα. Τις ανέφερε. Κάτι που σχετίζεται με τα κτίρια αλλά όχι με αυτό το συγκεκριμένο θέμα, αλλά θέλω να το πω. Είναι η ασφάλεια της πληροφορικής μας σε χώρες όπως η Κίνα. Θέλω μια ενημέρωση, δεν ξέρω αν γίνεται τώρα ή αργότερα για τα θέματα αυτά, γραπτός δηλαδή. Γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Θέλω ενημέρωση. Ο κύριος Κούς. Ευχαριστώ πολύ να επανέλθω σε αυτό που είπε η κυρία Χολμάια. Αυτέ είναι οι σωστέ ερωτήσει. Και προηγουμένω για τον Μπελμόντ, για τα κτίρια στι Βρυξέλλες. Τα ίδια ερωτήματα θέτονται, τίθενται τώρα και για το Πεκίνο. Πώ είναι η κατάσταση τώρα. Έχουμε την πρόθεση να συγκατοικήσουμε με άλλους θεσμούς ή ενδεχομένως και με εθνικούς θεσμούς από κάποια κράτη-μέλη, να ελέγξουμε. Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε έτσι μια συνεργασία για το κτίριο αυτό. Δηλαδή κοινή χρήση. Γιατί πρόκειται για νέο κτίριο. Ποιος είναι ο προγραμματισμός και ε, πώς έχουν τα θέματα ακριβώς επί των ερωτήσεων της κυρίας Χολμάιερ. Ο κύριος Λάρσεν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για τη στήριξή σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και αν ξεχάσω κάτι είναι γιατί δεν θα θυμάμαι τις ερωτήσεις, όχι γιατί θέλω να κρύψω κάτι. Πρώτον, για την ε, ανανέωση. Με βάση τον κινέζικο νόμο, οι ανανεώσει μισθώσεων μπορούν να γίνουν μόνο για τέσσερα χρόνια. Έτσι μας είπανε. Εγώ δεν νομίζω ότι σε τέσσερα χρόνια, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, ότι σε τέσσερα χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί το νέο κτίριο. Ίσως θα χρειαστεί να γίνει περαιτέρω ανανέωση της μισθώσεως, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ε, έτσι είναι η κατάσταση, εφόσον ε, οι ανανεώσει μισθώσεων είναι μόνο έως τετραετή. Α, και έτσι έγινε και κατά την προηγούμενη ανανέωση της μισθώσεως, έγινε το 2016. Μόνο τετραετής μπορεί να είναι λοιπόν η μισθώση Συνολικό κόστο. Τι έχω εδώ. Συνολικό κόστος. 1,4 εκατομμύρια. Όχι, 1,2. Το χρόνο. Κοιτάξτε, πρόκειται για ανανέωση μισθώματος, παράταση. Είδαμε τι γίνεται όσον αφορά τις αυξήσεις στην αγορά. Ακόμη και με αυτή την αύξηση είμαστε κάτω από τις μέσες αυξήσεις για τέτοιου τύπου κτηρίων. Ανά θα πληρώσουμε 33,4 ευρώ το μήνα. Ενώ οι τιμές της αγοράς θα ήταν, είναι, είναι 36-34 και ίσως ε, να, σε μερικέ περιπτώσει να είναι και 40 ευρώ ανά τετραγωνικό ανά μήνα. Άρα καλό. Καλή είναι αυτή η πρόταση. Καλή τιμή. Παρά την αύξηση η ασφάλεια των συστημάτων πληροφορική. Ναι, εξαιρετικά σημαντικό. Και είναι ένα από τα δύσκολα θέματα. Γιατί είναι ένα τεράστιο κτίριο, ε, αυτό που κτίζουμε τώρα. Ερωτήσαμε και άλλους που έχουν ε, χτίσει πρόσφατα στο Πεκίνο. Ε, είναι, είναι δύσκολο το θέμα. Υπάρχουν περιορισμοί στο πόσο ξένο προσωπικό μπορείς να φέρεις Ορισμένα τμήματα του κτηρίου θα πρέπει να έχουν ε, χωριστή ε, ασφάλεια 100%. Αλλά θα είναι δύσκολο να ελέγχουμε πλήρως συνολικά την οικοδόμηση αυτή. Γιατί αν κάναμε κάτι τέτοιο θα έπρεπε να αυξηθεί τρομερά το κόστος. Γιατί θα έπρεπε να πάμε εκεί πολύ επιπλέον προσωπικό. Αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό, απόλυτα σημαντικό θα επανέλθουμε από αυτού και με χαρά να το συζητήσω μαζί σας περαιτέρω. Αλλά είναι νωρίς ε, τώρα να πούμε τι θα κάνουμε. Θα επανέλθουμε. Τώρα κοινή χρήση και συνεργασία, συγκατοίκηση δηλαδή σε αυτό το κτίριο με άλλες υπηρεσίες. Επανέρχομαι, είχα προσπαθήσει και να απαντήσω. Κοιτάξτε, οι συνενικίε είναι πολύ σημαντική. Έχουμε μια ολόκληρη υπηρεσία που ασχολείται με το να ψάχνει τις δυνατότητες συνενοικίασης. Έχουμε γύρω στις 50 και μόνο ένα τρίτο είναι με κράτη-μέλη. Τα δύο τρίτα είναι με άλλους θεσμού της Ένωσης. Το Κοινοβούλιο ε, είναι ένας ε, καλός ε, συστεγαζόμενος χρεώνουμε κάτι, αλλά μόνο για τα δικά μα διοικητικά έξοδα. Δεν κερδίζουμε τίποτα. Για το Πεκίνο έχουμε αυτή τη στιγμή τρει συστεγάσει. Όλοι με άλλου ε, ευρωπαϊκού θεσμού. Την Τράπεζα Επενδύσεων, την, τράπεζα, την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και την EU IPO. Ήδη λοιπόν τρει συστεγάσει. Φυσικά δεν αποφασίζουμε για τα άλλα θεσμικά όργανα, αλλά οι περισσότεροι όταν περνάμε σε νέα φάση της στέγασής μας, έρχονται και αυτοί μαζί μας. Δεν μπορούμε πάντα να προγραμματίζουμε επακριβώς τις ε, δαπάνες μας, γι' αυτό έχουμε κάποιο περιθώριο, που είναι δύσκολο. Λόγω των προβλέψεων του δημοσιονομικού κανονισμού, αλλά χρειαζόμαστε ένα περιθώριο. Καταλαβαίνω γιατί δεν μπορείτε να μας το δώσετε. Αλλά στις και συνεργασίες είναι πολύ σημαντικό για όλα μας τα γραφεία στο εξωτερικό και στην Κίνα. Ευχαριστούμε κύριε Χολμάιρ. Είστε πραγματικός διπλωμάτης. Ε, αποφεύγετε το ζήτημα του Κοινοβουλίου, καταπληκτικά μας λέτε για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Μια χαρά τα λέτε. Αλλά για το Κοινοβούλιο θα σας στείλουμε τη λίστα του Κοινοβουλίου για τη συνενικίαση και μας ότι δεν υπάρχει παραπάνω κόστος και για τους άλλους ε, απεσταλμένους και αντιπροσώπους δεν υπάρχουν άλλα επιπλέον ε, κόστος. Το, η λίστα αρνείστε να μας τη δώσετε ε, με την οποία θα θέλαμε να συνεργαστούμε και για τα κονδυλία νομίζω είμαστε εντάξει γιατί η αύξηση των 44,6% μεταξύ 2002 και 2020 έχουν ανέβει οι τιμές αγοράς για πάνω από 92%. Καλύτερα από την υπόλοιπη αγορά. Μιλάμε για 500.000 ε, είναι η φθηνότερη τιμή ενοικίας που μας προσφέρει η αγορά. Άλλα σχόλια. Η τελική απόφαση λοιπόν γι' αυτό θα ληφθεί στην επόμενη συνεδρία. Σας ευχαριστώ. Τελευταίο σημείο στην ημερησία διάταξή μας, ανταλλαγή απόψεων για την παρακολούθηση των ψηφίσματων του Κοινοβουλίου και τη πρόοδου του Συμβούλου για το πολιτισμό νομικό πλαίσιο και του ιδίου πόρου. Καλό θα ήταν να πούμε ότι οι προτάσει τη Φιλανδική Προεδρία που δημοσιεύτηκαν στι 5 Δεκεμβρίου είναι πολύ κάτω από τι προσδοκίε του Κοινοβουλίου όσον αφορά την ε, εκπλήρωση των δεσμεύσεων τη Ένωση για την επένδυση, την νεολαία, το κλίμα και την ασφάλεια. Οι δεσμεύσει τη Προέδρου τη Επιτροπή Ursula von der Leyen, από την οποία μάθαμε και περισσότερα νέα χθε, θα είναι αδύνατο να υλοποιηθούν. Το προτινόμενο επίπεδο 1,07% ε, είναι μια εξίσωση αδύνατη. Δεν θα μας επιτρέψει να καλύψουμε τις προσδοκίες των πολιτών. Η πρόταση αυτή δεν είναι παρά το πρώτο βήμα πολύ δύσκολων διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο και με το Κοινοβούλιο φυσικά το οποίο θα πρέπει να δώσει τη συνένεσή του και είναι πλήρης συνομοθέτης ε, επιτομιακών πτυχών και κράτους δικαίου. Επομένως να γίνουν πολλά λοιπόν, αυτό είναι βέβαιο. Κυρία Μάρκες, θέλετε να σχολιάσετε. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ καλό να μπορούμε να το συζητήσουμε σήμερα αυτό. Μετά την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου και το ψήφισμα που υιοθετήσαμε με ευρεία πλειοψηφία για να υποστηρίξουμε έκθεση που είχε εγκριθεί από το προηγούμενο κοινοβούλιο στην προηγούμενη θητεία του Πέρση. Είναι ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου που υποστήριζε αυτήν την έκθεση που είχε προηγηθεί κυρίως δίναμε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα του, ε, το οικολογικού του κλίματος. Ε, γι' αυτό η πράσινη πρωτοβουλία, η πράσινη συμφωνία είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να ενταχθεί στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αλλά μας μένει ένα άλλο το πρόβλημα, ένα ζήτημα. Η χρηματοδότηση αυτής της πράσινης συμφωνίας. Δηλαδή με ποιες διαδικασίες, με τι τρόπους θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι θα μας προτείνει. Χωρίς να χρειαστούν νέοι ε, δημοσιονομική πόροι. Είτε και μάλιστα δεν ξέρουμε με τι συγκεκριμένες πολιτικές θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τι επιπτώσει των κλιματικών αλλαγών, ούτε πια θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα η συνεισφορά του Ευρωκοινοβουλίου. Εμεί καταστήσαμε σαφέ ότι θέλουμε 22% του συνολικού πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου να αφοσιώνεται σε στόχου ε, καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. Ε, σε κάθε περίπτωση ε, δεν θα είναι τελευταία φορά που το συζητάμε αυτό εδώ στην Επιτροπή μας. Σίγουρα η διαπραγματευτική ομάδα, η συγγήτρια και ο συνάδελφος ε, Όλμπριχτ μαζί με την εισηγήτρια, καθώς και οι εισηγητές και συνεισηγητές, ο κύριος Φερνάντες και η κυρία Αγέρ, καθώς και ο συνάδελφος Άντρεσεν, Ράσμος Άντρεσεν, πάντοτε εργαστήκαμε ως ένα κοινό μέτωπο, διότι θέλαμε να συμπαραταχθούμε με αυτά που είχε εγκρίνει προηγουμένως και το Κοινοβούλιο και να βρισκόμαστε διαρκώς και σε συνεννόηση με τους άλλους εισηγητές των άλλων αρμόδιων, επιτροπών. Από την πλευρά του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου είχαμε στήριξη στην όλη μας προσπάθεια να συνεννοηθούμε εσωτερικώς, να έχουμε μια καλή εσωτερική επικοινωνία, αλλά και με τους εξωτερικούς μας συνομιλητές. Ιδίω σε όσου έχουν διοριστεί υπεύθυνοι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ξέρουμε ότι στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο πρόεδρο Σασόλη για άλλη μια φορά θα υπενθυμίσει και θα υπογραμμίσει τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οργανώσαμε συνεδριάσει της ομάδα επαφή με συμμετοχή του Πρόεδρου του Κοινοβουλίου. Ε, οργανώσαμε συνεδριάσεις με τη συμμετοχή ε, εισηγητών των εισηγητών των διαφόρων ε, επιτροπών που ασχολούνται με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και κοιτάζουμε να ε, συνδυαστούμε με τις διάφορες εξωτερικές απόψεις που ακόμα να υπάρχουν ώστε να είναι διαρκής επικοινωνία με τις υπεύθυνε ε, επιτροπές και τις υπεύθυνου κοινοβουλίου. Είναι πολύ σημαντικό ο διάλογο, γιατί στο Κοινοβούλιο έχουμε διπλή ευθύνη. Πρώτα απ' όλα να μπορέσουμε να εγκρίνουμε το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτή είναι μία διαδικασία. Και μία δεύτερη είναι η αρμοδιότητα τη συναπόφαση. Αυτή που έχει το Κοινοβούλιο για κάθε συγκεκριμένο πρόγραμμα, για κάθε δημοσιονομική γραμμή στην επόμενη συνεδρίαση της ε, ε, διάσκεψης των Προέδρων, του Προεδρείου συγκεκριμένα. Ε, θα συζητηθεί πάλι αυτό το θέμα για να δούμε τι συγκεκριμένη στρατηγική θα ακολουθήσει κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή, ο κάθε ε, εισηγητής, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό πάνω απ' όλα να διαφυλάξουμε μια θέση τουλάχιστον επαναδίπλωσης, ε, ε, αν χρειαστεί, που ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί, και δεν, φτάσει καμία, δεν υπάρξει καμία συμφωνία σε κανένα γύρο τριμερού διαλόγου και δεν υπάρξει καμία έκβαση, θετική έκβαση στην όλη διαδικασία έγκρισης του πολίτης δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτή λοιπόν θα φανεί, αυτό θα φανεί και στα όσα θα συζητηθούν στη διάσκεψη των Πρόεδρων την ερχόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Κυρία Αγέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, σε ό,τι αφορά τους ιδίους πόρους. Με καλύπτει ο συνάδελφος Φερνάντες, μεν. Η διαδικασία είναι αυτή που περιέγραψε η Μαργαρίδα. Τώρα για το διαπραγματευτικό κουτί, για την πρόταση που θα γίνει. Έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες σε σχέση με το κείμενο που μας προτάθηκε αρχικά και υπήρξαν παρόλα αυτά ανησυχίε από την πλευρά τη Φιλανδική Προεδρία. Όχι μόνο γιατί θέτει να αμφιβόλο κάποια κεκτημένα, διότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει πει ότι θέλει απλούστευση, ενώ η Φιλανδία προτείνει πλήρη διαγραφή. Ε, Πρόκειται για πραγματικά ανησυχητικό στοιχείο και έπειτα περιορίζεται στο να ξαναδούμε του ίδιου πόρου κάνοντας το εξή την κλασική συνεισφορά. Στις διάφορες συνεδριάσεις που είχαμε ταυτόχρονα με τη Φιλανδική Προεδρία στο πλαίσιο της ομάδας ε, των ομάδων επαφή. θυμίζω ότι το Ευρωκοινοβούλιο ήθελε να γίνουν ε, βήματα πρόοδου στο θέμα των ιδίων πόρων, όμως αυτό ακριβώ τα καθόριζε και το πώ θα ψηφίζαμε για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν έχει γίνει κάτι καινούριο ω προ τη διαδικασία και σε σχέση με αυτά που μόλι μα είπε η Μαργαρίδα, γιατί είμαστε διαρκώ σε συνεννόηση και σε στενή συνεργασία σε επίπεδο δημοτευτικών ομάδων. Περιμένουμε να κάνει κάποιο βήμα και το Συμβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλα σχόλια. Ο κύριος Μουρεσάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα από την πλευρά μου να στηρίξω τους εισηγητές. Η γραμμή που μόλις περιγράψανε είναι αυτή που και στην πράξη ισχύει. Αυτή είναι η θέση του Κοινοβουλίου και θα πρέπει να συνεχίζουμε να εξηγούμε στο Συμβούλιο ότι ε, είναι η θέση που ακριβώ είχαν αναλάβει με τι δεσμεύσει του και αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Επίση, το Συμβούλιο δεν πρέπει να περιμένει ότι αργότερα στη διαδικασία θα πετύχουν μεταξύ του εκείνη μια συμφωνία και εμεί θα εγκρίνουμε ή θα κυρώσουμε ό,τι αποφασίσουν στο παρελθόν. Πάντοτε ανέβαλε τι αποφάσει στο Συμβούλιο. Διότι οι πρωθυπουργοί ή οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πάντοτε γνώριζαν ότι θα αποκυψουμε στι πιέσει τη τελευταία στιγμή. Αυτό παρελθόν λειτουργούσε για το κοινοβούλιο ε, μπορούσε να πει ναι, ε, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει τώρα. Και τρίτη παρατηρήση τώρα. Ε, θέλουμε φρέσκους, νέα κονδύλια, νέους πόρους. Και αυτό το επιβεβαιώνουν οι συνάδελφοι στην προηγούμενη διαδικασία του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Είχε αποφασιστεί το 2013 εκείνο. Και εκ τότε προβλέψαμε πολλά νέα προγράμματα που δεν τα ξέραμε στην αρχή του Πουδουπού. Το ε, πρόγραμμα Juncker, ε, ε, το, η, η, παράταση του ΕΦΣΙ, ε, το πρόγραμμα Εύση για την Αφρική, το Ταμείο για τους Πρόσφυγες, ε, ο τίτλος 3 που είχαμε ελάχιστο μηδενικό περιθώριο για τα επόμενα χρόνια και δεν μπορούσαμε να βρούμε καμία απόκριση για καμιά κατάσταση κρίσης. Γι' αυτό λοιπόν η απέτησή μας για ευελιξία, όλες οι απαιτήσει του Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικές. Ε, ε, οι προηγούμενοι κανόνες του Πουδουπού ήταν σωστοί και το νέο μήνυμα προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι το προηγούμενο σχέδιο ή μάλλον η προηγούμενη πρόταση της προηγούμενης επιτροπής του Μαΐου 2018 ήταν πολύ χαμηλή ε, στις φιλοδοξίες της, ε, μακριά από τις ε, επιθυμίες και τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου, τις απαιτήσεις και τις εκκλήσεις κρατών μελών στο Συμβούλιο και δεν μπορεί η περιοχή σύγκλησης να είναι μεταξύ του 1% που ζητούν κάποια κάτι μέλη και αυτό που έλεγε το προηγούμενο, η προηγούμενη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα είχε νόημα τέτοιο προπολογισμό. Και επίση να πω για του ιδίου πόρου. Και αυτό πολύ σημαντικό και θα είναι η μόνη πηγή για να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των αναγκών και αυτό που είναι έτοιμο να βγάλει από την τσέπη του και να πληρώσει το Συμβούλιο. Αυτό ε, το είπαν ε, και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνάδελφος Αγέ οι Ήδη πόροι μπορεί να είναι ε, η μόνη λύση. Και η τελευταία μου παρατήρηση, Πρόεδρε, είναι η εξή. Ότι κάποιε χώρε που είναι βασικοί συνεισφέροντε ακούνε από την κοινή του γνώμη να του λέει στι κυβερνήσει δηλαδή ότι πρέπει να κοιτάζετε πώ ξοδεύεται το ευρωπαϊκό χρήμα, αυτό που δίνουμε στην Ευρώπη. Οδηγεί στο εξή ερώτημα οι κυβερνήσεις που να λάβουν υπόψη πόσα θα δίνουν. Το καταλαβαίνω αυτό. Όμω τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει πολλά εργαλεία και μέσα για να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει χρηστή διαχείριση του ευρωπαϊκού Διαπολογισμού. Μετά έχουμε το ε, γραφείο την υπηρεσία του, του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Μετά έχουμε όλου του κανόνε για το κράτο δικαίου. Μετά την απλούστευση ε, των γραφειοκρατικών διαδικασιών και μεταξύ και μεταξύ άλλων και τη εκταμείευση ποσών. Αυτό το λέω γιατί πρέπει να το πούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πρέπει να το πούμε στι χώρε που επιμένουν στο 1%, στο περιθώριο. Ε, ο ευρωπαϊκό προπολογισμό θα εκτελείται καλύτερα στο μέλλον. Εμεί εργαζόμαστε πολύ ε, σκληρά για το σκοπό αυτό και πρέπει να είναι γι' αυτό βέβαιοι. Επίση, όλε οι πρωτοβουλίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρασίνισμα, το λεγόμενο Ταμείο Μετάβαση. Θα υπάρχει πραγματική μετάβαση, αν είναι ε, αρκετή η πρικοδότηση και δεν έρχονται τα ποσά από τι τσέπε τι δικέ μα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένα ταμείο μεν τη δίκαιη μετάβαση, αλλά πρέπει να παραμένουμε ενωμένοι ώστε η πρόταση για το κλίμα να μην επηρεάσει άλλε προτάσει και προγράμματα ή προτεραιότητε τη Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά την παρέμβαση των εισηγητών και του κυρίου Μουρεσάν, πολύ λίγα έχω να προσθέσω. Παρ' όλα αυτά, θέλω να διευκρινίσω ορισμένα θέματα. Προφανώ δεν είναι καλή η πρόταση τη Φιλανδική Προεδρία ούτε τα ποσά που προτείνει, ούτε το περιεχόμενό τη. Ε, δεν έχουμε την ε, μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση, δεν είναι πολύ συγκεκριμένες ε, οι ιεραρχήσεις, ε, για παράδειγμα το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση και μόνο εν μέρη δέχεται τα αιτήματά μας για την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά τα είχαμε πει εμείς οι βουλευτές στην προεκλογική εκστρατεία, αλλά τα είπε και το Συμβούλιο μέσω των αποφάσεών του και το Συμβούλιο όταν ε, όρισε τους υποψηφίους για επιτρόπους, γιατί οι κυβερνήσεις πρότειναν τους επιτρόπους που επεκύρωσε το Κοινοβούλιο και οι επίτροποι αυτοί δεσμεύτηκαν στις ακροάσεις ενώπιόν μας να προωθήσουν πολλές πρωτοβουλίες. Καθόλου δεν ανταποκρίνεται αυτή η πρόταση με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν και όλοι οι θεσμοί και εμείς μεμονωμένα προσωπικά. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να λέμε το ένα εδώ και το άλλο αλλού. Κοιτάξτε, όταν συζητούσαμε το 2012 ήταν ε, πολύ διαφορετικές προτεραιότητες. Τώρα έχουμε αυτές τις προτεραιότητες και πολλές άλλες. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Δεν είναι δυνατόν με το ίδιο ύψος πιστώσεων να καλύψουμε αυτά που ζητούσαμε τότε και αυτά που είναι αναγκαία τώρα. Η μόνη λύση σε όλα αυτά, η μόνη δυνατότητα να ε, υπάρξει τετραγωνισμός του προϋπολογιστικού κύκλου είναι περισσότεροι ήδη πόροι. Βλέπω ότι στο κείμενο της Φιλανδικής Προεδρίας υπάρχει μια δυνατότητα, ένα μικρό άνοιγμα της πόρτας προς περισσότερους ίδιους πόρους. Πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Βλέπουμε τουλάχιστον κάποιο μικρό περιθώριο αισιοδοξία και Θέλουμε να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και τους επόμενους μήνες θα κάνουμε πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Ότι ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε χωρίς να ζητήσουμε περισσότερη χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη είναι περισσότερη ήδη πόροι. Κάτι άλλο που με ανισχύει ιδιαίτερα στα πλαίσια της ε, φιλαδικής προεδρίας, της πρότασής της, τα Nego Box, η, τα κουτιά διαπραγματεύσεων, έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με τη συναπόφαση να σας δώσω ένα παράδειγμα που είναι δικό μου θέμα. Το πρόγραμμα στήριξης στις ε, μεταρρυθμίσεις. Το Κοινοβούλιο ούτε έκθεση δεν μπορούσε να κάνει. Γιατί η πρόταση της Φιναλικής Προεδρίας είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θέλουμε. Έχουν ήδη όλα αποφασιστεί. Έχουν αποφασίσει πόσα θα είναι, τα κριτήρια για την κατανομή, πώς θα ληφθούν οι αποφάσεις, όλα έχουν ήδη αποφασιστεί. Τα έκαναν όλα. Και είναι όλα εκεί πέρα μέσα σε αυτό το Nego Box. Κοιτάξτε. Υπάρχουν πολλές παρόμοιες λεπτομέρειες και για τη συνοχή και για τη γεωργία. Αυτά δεν είναι νόμιμα. Δεν είναι ε, κανονικά με βάση το πλαίσιο των διοργανικών ε, σχέσεων. Πώς είναι δυνατόν ε, να προκαταλαμβάνονται τέτοια πράγματα. Έχουμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις ακόμη. Γιατί θα είναι δύο αποφάσεις που θα ληφθούν με συναπόφαση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ανδρέης. Ευχαριστώ. Οι διαπραγματεύσεις για το δημοσιονομικό πλαίσιο κυρίως πρέπει να δουν ε, προς ποια κατεύθυνση θα πάμε. Όμως τώρα συζητάμε για λεπτομέρειες, ε, κάνουμε παζάρια και κάποιες πλούσιες χώρες όπως η Ομοσπονδιακή Γερμανία δεν βοηθάνε. Μπλοκάρουν τη διαδικασία. Ανησυχητικό πολύ αυτό. Θα έπρεπε να είμαστε σε άλλο σημείο τώρα. Έγιναν κάποιες πρόοδοι τους τελευταίους μήνες, αλλά είναι ανεπαρκείς. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να συζητάμε λεπτομέρειε μόνο. Συζητήσαμε χθε για την πράσινη συμφωνία στην Ολομέλεια. Εκεί είμαστε, είπε η Φοντελάιν. Αλλά σήμερα τα κράτη-μέλη επίσης φαίνεται ότι θα αποφασίσουν ότι μέχρι το 2050 θα πρέπει να είμαστε κλιματικά ουδέτεροι. Αλλά μετά στο δημοσιομικό πλαίσιο δεν κάνουμε τα αντίστοιχα. Εδώ είναι το βασικό θέμα. Διότι τα νούμερα έτσι όπως είναι τώρα δεν αρκούν καθόλου για να επιτύχουμε τους κλιματικούς μας στόχους. Για να είμαστε κλιματικά ουδέτεροι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Και οι προτάσεις της Κομισιόν, οι χθεσινές, υπευλήθησαν και άμα δει κανείς ακριβώς τα ποσά για τα θέματα του κλίματος είναι τα παλιά στοιχεία. Χρειαζόμαστε νέα στοιχεία, νέες προτάσεις για την πράσινη συμφωνία. Πρέπει να ενταχθεί στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Και όχι κατόπιν κάποια στιγμή όταν θα επιτύχουμε συμβιβασμό για το δημοσιονομικό πλαίσιο τότε να δούμε πώ με κάποιο τρόπο θα έχουμε ένα σχέδιο επενδύσεων για την πράσινη συμφωνία. Γι' αυτό θα ήθελα σήμερα να έχουμε εδώ τον Επίτροπο. Για τα θέματα αυτά δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα κράτη-μέλη, έχουν να κάνουν και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να συζητηθούν. Ξέρουμε, για παράδειγμα, από το ελεγκτικό συνέδριο ότι θα χρειαστούμε 1,2 δις το χρόνο στα πλαίσια του δημοσιονομικού πλαισίου δεν προβλέπεται. Και επίσης έχουμε και χρονικά καθυστέρηση. Όσο τα κράτη-μέλη τσακώνονται και δεν καταλήγουν σε συμφωνία, καθυστερούμε. Γιατί θα ξεκινήσουν κατόπιν τα προγράμματα αργότερα. Αυτό έχει να κάνει και με τη χρηματοδότηση τη γεωργία μα, τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, με όλου του δικαιούχου που περιμένουν χρηματοδοτήσει από εμά. Είναι σημαντικό επιτέλου το Συμβούλιο να σηκώσει τα μανίκια του, να κάνει κάτι. Τσακώνονται εδώ και εβδομάδε και δεν έχουν αλλάξει οι όροι του τσακωμού. Πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση και να επιτύχουμε συμφωνία για τους στόχους της κλιματικής ουδετερότητας. Χαίρομαι που στο τέλος μπορώ να πω ότι υπάρχει ομοφωνία στην διαπραγματική ομάδα του Κοινοβουλίου και κάνουμε κάθε προσπάθεια να επιτύχουμε καλού συμβασμού. Και του επόμενου μήνε πρέπει να ενημερώσουμε περισσότερο την κοινή γνώμη γι' αυτό και να καταδείξουμε τα κράτη-μέλη. Αυτά πρέπει να μετακινηθούν για να υπάρξει συμφωνία. Έτσι θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε την κοινή γνώμη που ίσως είναι επικριτική σε ορισμένα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και πρέπει επιτέλους το Συμβούλιο να μετακινηθεί για να επιτύχουμε κάποια συμφωνία. Ευχαριστώ. Ο κ. Παπαδημούλης. σημειώνω ως ιδιαίτερα θετικό ότι όλες οι πολιτικές ομάδες απορρίπτουν κατηγορηματικά την πρόταση της Φιλανδικής Προεδρίας και νομίζω ότι το κάνουμε γιατί έχουμε συνεννοηθεί ότι για να χρηματοδοτηθούν οι πολιτικές και οι στόχοι που έχει δει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που έχει δει ακόμη και η Κομισιόν, η οποία προέκυψε μετά από προτάσεις των κυβερνήσεων, η πρόταση που έχουμε καταθέσει ως Κοινοβούλιο εδώ και ένα χρόνο είναι απολύτως απαραίτητη, το 1,3% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η δήλωση που θα κάνει ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ο κύριος Σασόλη, σε λίγες ώρες ε, στο Συμβούλιο απορρίπτοντας κατηγορηματικά την πρόταση της Φιλανδικής Προεδρίας και ζητώντας έναν πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό. Θεωρώ επίσης σημαντικό ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ανεξάρτητα από τις διαφορές μας, υπερασπίζουμε ε, το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που λέει ότι το 1,3% είναι απολύτως απαραίτητο για να χρηματοδοτηθούν όσα ζητούν οι πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση της Φιλανδικής Προεδρίας νομίζω ότι προσβάλλει και την κοινή λογική και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ως συνομοθέτης πρέπει να διεκδικήσει το ρόλο του, για να μην υποστούμε ταπεινωτική μεταχείριση στο όνομα του επίγοντος, με το επιχείρημα ότι ο χρόνος τρέχει και πρέπει να κάνουμε μεγάλες υποχωρήσεις η φιλανδική πρόταση μειώνει την πρόταση του Κοινοβουλίου κατά 13% για την περιφερειακή ανάπτυξη, κατά 27% για την κοινωνική συνοχή, κατά 25% για το πρόγραμμα LIFE για το κλίμα, κατά 30% για το πρόγραμμα Horizon, κατά 48% για το πρόγραμμα Εράσμους, κατά 35% για το πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη. Και την ίδια ώρα, αν συγκρίνουμε την πρόταση της Φιλανδικής Προεδρίας με το προηγούμενο MFF, αυτό που ολοκληρώνεται, προβλέπει αύξηση 132% για τη διαχείριση των συνόρων και τη μετανάστευση και 650% για την ασφάλεια και την άμυνα. Πώς μπορούμε αυτά να τα δικαιολογήσουμε στους πολίτες. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι λυπηρή η απουσία του Επιτρόπου Χάν σήμερα από την Επιτροπή μας θα έπρεπε να είναι εδώ ο νέος Επίτροπος για να δείξει μια διάθεση επικοινωνίας και συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμφωνώ και με όσους συναδέλφους είπαν ότι πρέπει να πιέσουμε για να αυξηθούν, να ενισχυθούν οι ίδιοι πόροι. Ο μόνος τρόπος να σταματήσουν να τσακώνονται αδιεξόδως οι net contributors και οι net receivers στο Συμβούλιο, οδηγώντας διαρκώς προ τα κάτω το, το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι να αυξηθούν οι ίδιοι οι πόροι. Και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πιέσει οι προτάσει τη Επιτροπής Μόντι να βγουν από το σιρτάρι, να τεθούν στο τραπέζι της συζήτηση και πάνω εκεί να επιδιώξουμε τις πιο φιλόδοξε λύσει. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Κύριε Κορμό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ανταλλαγή απόψεων αυτή. Τώρα, για να είμαι ειλικρινή, ε, πέραν τη απόλαυση αυτή τη ανταλλαγή απόψεων, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει όλη αυτή η συζήτηση, αφού τελικά θα μιλήσει ο Επίτροπο. Οπότε... Και αφού δεν είναι εδώ, τι συζητάμε. Η προσέγγιση για αυτό το πολιτιστικο δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ότι πρέπει να βασιστούμε σε νέα πολιτικά ε, δεδομένα. Άκουσα την πρόεδρο χθε ε, και πολύ μιλήσαμε εδώ σήμερα για αυτό το Green Deal, το Πρασινό Σύμφωνο. Τη δεκαετία του 30 είχαμε το New Deal στην Αμερική, και σήμερα αυτό μας ενέπνευσε για να μιλήσουμε τώρα Green New Deal. Σήμερα τότε υπήρχε μια οικονομική κρίση και ο πρώτος Ρούσβελτ αύξησε τη φορολογία τη δεκαετία του 30. Χρεώθηκε. Ξεκίνησε μια μαζική πολιτική επενδύσεων με στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη. Για να φτιάξουμε εμείς ένα Green Deal σήμερα δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε αν εξακολουθήσουμε να ακολουθούμε την ίδια προσέγγιση με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μένα λοιπόν σε αυτή την υπόθεση είναι ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τον προπολογισμό και θα είναι περίπλοκο αυτό με τα κράτη-μέλη και ειλικρινά αν είμαστε στο 1,1613. 13 ούτως ή άλλως δεν καλύπτουμε τις ανάγκες μας οπότε το βασικότερο διακύβευμα για να αλλάξουμε προσέγγιση είναι το ζήτημα των ιδίων πόρων για να αλλάξουμε κλίμακα. Και με ανησυχεί εδώ η, πρόταση της Φιλανδικής Προεδρίας. Γιατί φυσικά ανοίγει μια πόρτα, ε, θεωρούμε ότι η πόρτα είναι ανοιχτή γιατί δεν την έκλεισε κανένας, αλλά εγώ θεωρώ ότι μας πάει πίσω η πρόταση αυτή. Ε, το ΦΠΑ που ήταν ένας ιδιοσπόρος ατελής αλλά που υπήρχε και για τους άλλους ε, νέους ιδιοσπόρους που προβλέπονται ο φόρος για τα πλαστικά είναι η μόνη που φαίνεται να αξίζει κάτι, αλλά δεν έχουμε την πλήρη πρόταση ακόμα και αλλιώς δεν υπάρχει τίποτα και από ό,τι κατάλαβα ε, το φόρο για την κυροζήνη ούτε το συζητάμε. Κρίμα, διότι θα ήταν εύκολος ε, φόρος στην εφαρμογή του και πολύ δίκαιος ε, κοινωνικά, γιατί οι Ευρωπαίοι πολίτες όταν βάζουν βενζίνη στα αυτοκίνητά τους φορολογούνται, αλλά όταν ε, βάζουμε καύσιμα στα αεροσκάφη, εκεί δεν φορολογείται κανεί. Οπότε είναι αναγκαίο να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το ζήτημα. Θέλουμε μεγαλύτερη αυτονομία δημοσιονομική ω κοινοβούλιο, ούτω ώστε να υπάρξει μια φορολογία ε, πιο οικολογική και που θα μας δώσει και ίδιους πόρους αρκετούς για τις εποχές που έρχονται. Τώρα, υπάρχει και άλλο ένα θέμα που θα ήθελα να συζητήσουμε μεταξύ μας Αφού έχουμε την ευκαιρία θα ήθελα να μάθω σε ποιο βαθμό θα συνεχίσουμε να συμφωνούμε όλοι μαζί μέχρι το τέλος γιατί η θέση του Κοινοβουλίου ήταν ισχυρή, ήμασταν όλοι ενωμένοι. Θέλω να μου πείτε, δώσαμε κάποια ένδειξη μέχρι πού θα το πάμε σε αυτό το μπραντεφέρ με το Συμβούλιο. Ε, δεν θα δεχθούμε τις προθεσμίες που πάνε να μας επιβάλλουν θα δεχθούμε να τραβήξουμε τα πράγματα στα άκρα εάν δεν καταφέρουμε να επιτύχουμε αυτό που θέλουμε. Διότι όσο και να συζητάμε μεταξύ μας έχουμε απαιτήσει, έχουμε απαιτήσει και μετά ξαφνικά πάμε ε, και συζητάμε και τελικά στο, σε θέματα χρονοδιαγράμματος ε, συμφωνούμε, δεν έχει νόημα όλο αυτό. Πόσο μάλλον θα μας αποδυναμώσει τελικά. Εάν λοιπόν ε, δεν καταφέρουμε να ε, συνεφέρουμε κάποιο στο Συμβούλιο, θα πρέπει να επιμείνουμε, να τραβήξουμε τα πράγματα στα άκρα, να μην ε, για να προβληθεί αυτό και στην κοινή γνώμη. Δεν είμαι βέβαιος ότι η κοινή γνώμη θα αντιτεθεί σε αυτό που προτείνουμε εμείς και θα υποστηρίξει αυτό που προτείνουν τα κράτη. Οπότε πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση μεταξύ μα για να δούμε μέχρι πού σκοπεύουμε να το πάμε. Χρονικά δηλαδή. Ευχαριστούμε. Κύριε Κόνα. Θα μιλήσω γερμανικά. Είπε ήδη ο Πρόεδρος να είμαστε σύντομοι και θα είμαι σύντομος. Αντιλαμβάνομαι όσα συζητάμε, πόσο συχνά συζητάμε εδώ στην Επιτροπή αλλά και στη διαπραγματευτική ομάδα, στην ομάδα επαφής του Κοινοβουλίου και η θέση μας είναι σαφέστατη. Έχει έρθει η ώρα να μετακινηθούν λίγο και τα κράτη-μέλη. Θέλω να υπογραμμίσω ένα θέμα από αυτά που είπε ο συνάδελφος Μοροζάν. Είναι σημαντικό, πιστεύω, ειδικότερα στις χώρες που συμμετέχουν ε, σημαντικά στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί τους απασχολεί το θέμα αν θα υπάρχει λογική διαχείριση των δαπανών. Ε, δεν είναι 100% βέβαιο στο negotiating box των Φιλανδών δεν είναι βέβαιο ότι θα επιτευχθεί η ε, ειδική πλειοψηφία που απαιτείται. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς ως κοινοβούλιο για μας είναι σημαντικό καθοριστικό σημείο. Το πόσο μεγάλη θα είναι η αποδοχή μεταξύ των πολιτών θα πρέπει να την ενισχύσουμε αυτήν. Οπότε θα πρέπει να κάνει περισσότερες προσπάθειες στο κοινοβούλιο. Ε, να παγιωθεί και αυτός ο μηχανισμός του κράτους δικαίου. Πιστεύω θα πρέπει να υπερασπίσουμε περαιτέρω την ισχυρή θέση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε κύριε Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τρία πράγματα έχω να πω. Πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι η γλώσσα που χρησιμοποιούμε δεν πρέπει να δείχνει ότι είμαστε σε ρήξη με τα κράτη-μέλη. Ω κράτη-μέλη ξεκινάμε από διαφορετική αφετηρία για να επιτύχουμε του στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και οι διαφορετικέ αυτέ αφετηρίες σημαίνουν ότι υπάρχουν διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών. Η Πολωνία, για παράδειγμα, δεν έχει λόγο να διαμαρτύρεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε εγώ έχω τέτοιου λόγου. Αλλά θα πρέπει να πούμε στου Ευρωπαίου πολίτε, καθαρά ότι ξεκινάμε από διαφορετικέ αφετηρίε. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του νέου Πράσινου Συμφώνου, το νέο, το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι λαμβάνοντας υπόψη το σχεδόν ιστερικό αφήγημα για το Πράσινο Σύμφωνο και για τους στόχους που έχουμε θέσει αλλά τα χρήματα που δεν υπάρχουν για να τους επιτύχουμε. Το να πάρουμε για παράδειγμα χρήματα από το Μηχανισμό σύνδετα στην Ευρώπη ή από άλλες πολιτικές για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς ε, πιθανότατα να μην είναι η καλύτερη λύση που θα μπορούσαμε να επιλέξουμε. Θυμηθείτε, η Ευρώπη δεν είναι σαν τον υπόλοιπο κόσμο και ο υπόλοιπο κόσμο δεν είναι σαν την Ευρώπη. Όταν πάω και βλέπω τι κάνει η Κομισιόν και τι κάνει το Κοινοβούλιο, το βλέπω στο πλαίσιο του ανταγωνισμού μας με τις άλλες οικονομίες. Βάσει αυτού θα διαμορφώσουν άποψη στο μέλλον οι ψηφοφόροι μας. Κατά πόσο θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και αυτό πιστεύω θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα, ειδικότερα να δούμε τον ενεργειακό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο και των υπόλοιπων πολιτικών που υλοποιούνται στην Κίνα, στην ε, υπόλοιπη Ασία, στη ΣΥΠΑ. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και για να κλείσω, η φιλανδική πρόταση δεν μας οδηγεί πιο κοντά σε συμβιβασμό. Θα ήθελα να μην χαλάσουμε τις σχέσεις μας και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις νέες προκλήσεις βάσει της φιλανδικής ε, πρότασης. Η Πολωνία είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί κατανοούμε τους στόχους, αλλά χρειαζόμαστε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τις διαπραγματεύσεις μας στο πλαίσιο του πολιτισμού νομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Σφάτσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να του ζητήσω να εστιαστεί σε δύο ζητήματα. Πρώτον, ποια είναι η αξιολόγηση της Κομισιόν όσον αφορά τα, μόλις, ε, τα όσα μόλις πρότεινε η Φιλανδική Προεδρία και δεύτερον, ποια θα είναι η θέση που θα ε, λάβει σήμερα ο Επίτροπος στις συζήτηση που θα γίνουν αργότερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί εισηγητέ, ευρωβουλευτέ, συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ο Επίτροπο Χάν ζητά συγγνώμη. Δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ, διότι έχει λυμμένε υποχρεώσει. Όμω είναι διατεθειμένο να συνεργαστείτε στενά, όπω συνέβαινε και την περασμένη δεκαετία όσο ήταν Επίτροπο. Ε, με τα χαράς να απαντήσω στα ζητήματα, στα σημεία που έθεσε μόλις ο Πρόεδρος. Όπως όλοι γνωρίζετε, η Φινλανδική Προεδρία υπέβαλε μια πρόταση που ονομάζεται Negotiation Box, διαπραγματευτικό κουτί. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το βλέπει σχετικά θετικά, το Κοινοβούλιο πολύ επικριτικά. Κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα δούμε λίγο διαφορετικά, γιατί ίσω και να είναι επικοδομητικά στο έγγραφο αυτό και κάποια που τα βλέπουμε πολύ αρνητικά ή πολύ, ιδιαίτερα αρνητικά. Στα θετικά, η ευθυγράμμιση των σκοπών του κλίματος με πρικοδότηση 25% βρίσκεται στο κουτί και είναι εντό αγγυλών μεν, αλλά ένα πολύ καλό βήμα για το μηχανισμό κράτους δικαίου. Έχουμε πλέον ένα κείμενο στο έγγραφο που είναι πολύ κοντά στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επίσης αναφερόταν στο κράτος δικαίου κάτι που είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως η αντιστραμμένη ενισχυμένη πλειοψηφία βρίσκεται εντό αγγυλών, αλλά θα καταλαβαίνετε όλοι ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα λεπτό και θα κρυθεί στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ε, σημαντικά στοιχεία είναι τα ποιοτικά στην πολιτική συνοχή, η θεματική συγκέντρωση, οι μεταφορέ στη συνοχή. Κάποιες από τις εφαρμοστικές ε, διαδικασίες είναι θετικό ότι θα υπάρχει ένταξη στον προπολογισμό του ETF και ε, δεν θα υπάρχει εργαλείο για τη γειτονία όπω συνέβαινε στο προηγούμενο διαπραγματευτικό κουτί. Αυτά είναι βήματα προόδου και νομίζω ότι τα εκτιμά θετικά και το Κοινοβούλιο. Και σωστά υπάρχει και αναφορά στο Ταμείο Δίκαιη Μετάβαση και στο Μηχανισμό Δίκαιη Μετάβαση. Όπω είπαμε, περιμένουμε ε, νομική πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι 14 Ιανουαρίου, για το θέμα αυτό. Στα αρνητικά πρώτα απ' όλα. Βεβαίω, στο συνολικό επίπεδο το 1,7%. Στο 1,07%. Θεωρούμε ότι ο τρόπος που γίνεται ε, αυτό είναι ότι όλες οι ενισχυμένες προτεραιότητες, Frontex, Ταμείο για την Άμυνα, προγράμματα για την ανταγωνιστικότητα, όλα αυτά μειώνονται. Ε, τα εξωτερικά προγράμματα περιορίζονται. Όλες αυτές οι περικοπές ε, είναι 47 εκατομμύρια ευρώ και θεωρούμε ότι οι περικοπές αυτές, μετά μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, δημιουργούν προβλήματα. Αυτό η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ελπίζουμε, δεν είναι πλέον προτινόμενη, έχει εκλεγεί, ελπίζουμε θα τα πει και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα τα ξεκαθαρίσει. Ένα άλλο θέμα είναι οι περικοπές στα διοικητικά στη δίκηση. Άκουσα με ενδιαφέρον τη συζήτηση για τον προπολογισμό και την κτηριακή πολιτική προηγουμένω. Οι περικοπέ στα διοικητικά είναι 2 δι ευρώ. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του προσωπικού όλων των θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωκοινοβούλιο αυτό, αν αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα το οποίο σας προβληματίζει και για το οποίο θέλετε να αγωνιστείτε και να το ε, κυρώσουμε. Για τους νέους ιδίους πόρους. Θα πρέπει να συμφωνήσω με αυτό που είπε η κυρία Γκαρδιαθαμπάλ. Ε, είναι ανεπαρκές αυτό που προτείνεται στη φιλανδική πρόταση στο κουτί. Βεβαίω υπάρχει κάποια πρόοδο. Δηλαδή η συνεισφορά με το φόρο των πλαστικών εντό αγγυλών, έστω μια νέα δημοσιονομική γραμμή για άλλου ενδεχόμενου νέου πόρου και αυτό εξαιτία τη πίεση του Ευρωκοινοβουλίου που εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καλωσορίζουμε. Ελπίζουμε να συνεχίσετε να ασκείτε πίεση ε, στα προσυπόμνηση ε, των ιδίων πόρων. Λοιπόν. Ε, τώρα για την ευελιξία. Ίσως δεν έχει υπογραμμιστεί αρκετά. Θεωρούμε ότι όσα περιλαμβάνει η πρόταση είναι σοβαρότατη μείωση και περιορισμό τη ευελιξία. Θα θυμάστε όλοι το πρόβλημα του backlog που είχαμε το 2014 και εφ' Έχουμε δυστυχώς μειώσουν τι δυνατότητε μας να αντιμετωπίζουμε τέτοια θέματα και πραγματικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι λίγο υπόγειο ε, όλοι μιλάνε για τα μεγάλα και τα πιο ορατά, όμω ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να πιέζει όπω κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι το επίπεδο ευελιξία ε, στην πραγματικότητα ε, επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βρίσκει κάποια απόκριση σε κρίσει, όπω κάναμε με το τωρινό δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τουλάχιστον το σημερινό επίπεδο το κείμενο της πρότασης της Φινλανδικής Προεδρίας είναι κάτω από το επίπεδο της ευελιξίας που έχουμε σήμερα. Είναι σαφές αυτό, το βλέπουμε ιδιαίτερα αρνητικά αυτό το σημείο. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να τα δούμε στην επόμενη διαπραγματευτική φάση του λεγόμενου διαπραγματευτικού κουτιού. Το επόμενο βήμα είναι ότι θα αναλάβει η επόμενη Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εμεί ενθαρρύνουμε και αυτό είναι ένα άλλο μήνυμα που θα περάσει απόψε από την Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι να περάσουμε σε μια γοργή συμφωνία για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε καθυστερήσει ήδη πάρα πολύ. Ξέρετε ότι την προηγούμενη φορά είχαμε ήδη καθυστερήσει για την αρχή υλοποίηση των προγραμμάτων και θεωρούμε και αυτό ίσως έχει παραβλεφθεί κάπως. Ο διάλογος με το Ευρωκοινοβούλιο της κρατικής προεδρίας πρέπει να προχωρήσει ε, με την Προεδρία του Ευρωκοινοβουλίου. Θα πρέπει το Συμβούλιο να γνωρίζει επακριβώς ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, έχουμε συστηματικά διάλογο και επικοινωνία μαζί τους. Ε, ενθαρρύνουμε και προτρέπουμε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή είναι η δική μου ανακεφαλαίωση. Η ανακεφαλαίωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα βασικά σχόλια ε, που θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ ε, για να εκφράσω τι απόψει τη Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Φιλανδική Προεδρία. Κυρία Μάρκε, για τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, καταρχά να ευχαριστήσω όλου για τι συνεισφορέ του και όλε οι παρατηρήσει ήταν χρήσιμε. Πράγματι, είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργήσουμε αυτό το διάλογο και έχουμε εντοπίσει Δεν έχετε μετάφραση, ρωτάει η ομιλήτρια. Ωραία. Ε, ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις παρατηρήσεις που έκανε, γιατί είναι και για μας πραγματικά αυτά σημαντικά. Είναι προτεραιότητες που τις είχε θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όπου θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Σε ό,τι αφορά το διαπραγματευτικό κουτί, είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι σε αυτή τη φάση τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου γνωρίζουν επακριβώ τι θέσει του Ευρωκοινοβουλίου. Δηλαδή, το Κοινοβούλιο απέστειλε στη Φινλανδική Προεδρία και στην ε, Υπουργό του Πουράινεν, που τα μοίρασε σε όλα τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, την απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο δημοτευτικό κουτί. Όλοι οι υπουργοί γνωρίζουν αυτή τη στιγμή τι θέσει του Κοινοβουλίου για καθένα από τα σημεία ξεχωριστά. Και αυτό, κατά την άποψή μου, είναι ε, ιδιαίτερα σημαντικό για να προσπαθήσουμε να βγούμε από τη δύσκολη θέση. Ω προ το διάλογο τουλάχιστον το διαθεσμικό για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Για τα σημεία που θίξατε ω προ του πολίτε και την κοινή γνώμη. Η εικόνα που έχουν διαμορφώσει οι πολίτε για το πώ χρηματοδοτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πιστήσω την προσοχή σα στην προσπάθεια που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το να δημοσιοποιήσει αριθμούς λόγου χάρη για το κέρδος που προκύπτει την εσωτερική αγορά. Αλλά να θυμίσουμε και τη διάσταση που ο Γιωχάνης Χάν επεσήμανε εδώ ε, σε μια προηγούμενη παρέμβασή του στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή ότι δεν μπορούμε να μείνουμε ε, στην ε, ιεράρχηση των των χωρών που συνεισφέρουν ε, ξεκάθαρα και ε, αυτόν που είναι απλώς δικαιούχοι. Ε, δεν μπορεί να μείνει η ιεράρχηση του παρελθόντος. Δεν είναι αυτό σωστή εικόνα για να δίνουμε στους πολίτες των κρατών και πρέπει να έχουμε μια επικοινωνιακή στρατηγική ώστε να καταλαβαίνουν οι πολίτες ακριβώς ποια είναι τα ωφέλη που αποκομίζουν η προσθεθέμενη αξία και η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ' επέκταση του προπολογισμού της. Ε, έγινε μια παρατήρηση επίσης, πολλές παρατηρήσεις για τους ιδίους πόρους. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε το μέλλον και να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, εάν δεν υπάρξει προηγουμένως σαφήνεια και πραγματικά ε, επιμένω στον όρο σαφήνεια, όχι απόφαση, σαφήνεια για τους ιδίους πόρους. Ε, πραγματικά ο προπολογισμό όπως χρηματοδοτείται σήμερα με το υψηλότερο ποσοστό να καλύπτεται από το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του κάθε κράτου μέλου, ε, θα μα οδηγεί κάθε φορά να ακούμε τα ίδια και τα ίδια και τελικά να μην έχουμε ποτέ έναν επαρκή προπολογισμό για να χρηματοδοτήσουμε τι προτεραιότητε τη Ένωση. Τέλο. για την μελλοντική προεδρία και τη, τη δική μας διαπραγματευτική ομάδα ε, πρέπει να πω ότι έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με του εκπροσώπους της κρατικής Προεδρίας και θα έχουμε διμερεί συνομιλίε μαζί τους. Ε, και εφόσον χρειαστεί και με τη Γερμανική Προεδρία θα πρέπει να είμαστε ε, ξεκάθαροι και σαφείς στη στατικική μας για το τι θα κάνουμε με τις δύο προεδρίες που επίκυνται. μετά τους Γερμανούς έχουμε Πορτογαλική Προεδρία. Ε, κάτι πολύ σημαντικό επίσης και ένα θέμα που να το θέσω οπωσδήποτε εδώ, ιδίω μετά την παρέμβαση του Ράσμους. Όλες οι πολιτικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να χρηματοδοτούνται εντός προπολογισμού και βάσει των κανόνων του. Δηλαδή να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια και πράγματι το ε, ε, Ευρωκοινοβούλιο να διαδραματίζει το ρόλο που το αναλογεί. Δεν μπορούμε να βρισκόμαστε σε καταστάσεις όπως αυτή που επίκειται ίσως να δεχτούμε για να βγούμε από τη δύσκολη θέση των δημοτεύσεων του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου να χρηματοδοτούμε πολιτικέ πρωτοβουλίε εκτό προπολογισμού, εκτό κουδουπού. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί προ αυτό και πολύ προσεκτικοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνω τη συζήτηση για το θέμα αυτό και η συνεδρίαση τη επιτροπή μα. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα είναι στο Στρασβούργο 13 Ιανουαρίου θα είναι κοινή Badge Econ με τον κύριο Χόιερ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και η επόμενη συνεδρίασή μας στις Βρυξέλλες θα είναι 22-23 Ιανουαρίου, όπου, όπως ε, άτυπα μόλις ακούσαμε, θα έχουμε τον κύριο Χάν. Ευχαριστώ πολύ.